ιστοσελίδα της Ολομέλειας. Ε, ε, το επόμενο δεν ξέρω αν είναι σωστό για τις επενδύσεις παιδιά Αντώνιο Λόπες Ιστορίστσε και 10 ε, ακόμη συγκέντρωσε 458 υπογραφές και έχει την πλειοψηφία με βάση το άρθρο 36 του κανονισμού η δήλωση αυτή μαζί με τα ονόματα των υπογραφόντων θα δημοσιευθούν και θα σταλούν ε, στους